Εσύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη σκληρή δουλειά σας, τη συμβολή σας. Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και όλους τους βουλευτές, καθώς και, όλους, ε, και για όλους όσοι επιστρέφετε